Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Euh, Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον κύριο Μίλη και τον συγχαίρω για την παράταση της θητείας του, γιατί τώρα είναι επέκταση μάλλον, Γενικός Διευθυντής από την 1η Σεπτεμβρίου ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και όχι πλέον εκτελεστικός διευθυντής. Ανέκαθεν συνεργαζόσαστε με την Επιτροπή και στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου μας παρουσιάσετε και το πρόγραμμα των εργασιών σας. Με χαρά θα σας ακούσουμε να μας παρουσιάσετε το όραμά σας για το μέλλον γιατί είστε πλέον γενικός διευθυντής αυτού του περίφημου οργανισμού. Σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις νέες σας προτάσεις και τους προσανατολισμούς για το μέλλον. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους παρόντες ευρωβουλευτές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου και πάλι να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην Επιτροπή σας που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητες του οργανισμού και την επέκταση ε, της εντολής μου ως εκτελεστικού διευθυντή. Έχουμε συνεχή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι ύψης της σημασίας αυτό για ε, τον οργανισμό μας και το προσωπικό του. Όταν ήρθα τον Ιανουάριο ενώπιόν σας, σας έδειξα την παρούσα διαφάνεια που τονίζουμε τις ε, προτεραιότητες και τις προκλήσεις για το 2017. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στη νέα συνεργασία για την ακτοφυλακή που ε, είναι καθοδόν ακόμα αυτή η αποστολή μας. Τώρα προσλαμβάνουμε προσωπικό με τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα για να ανταποκριθούμε στο έργο μας και στην εντολή μας και συντονίζουμε τις δραστηριότητές μας. Η πρόσφατη μεταναστευτική κρίση οδήγησε σε έντονη νομοθετική δραστηριότητα αλλά και σε μεγαλύτερη εστίαση για τις δραστηριότητες του λιμενικού σώματος και της ακτοφυλακής. Στην εντολή μας, ε, όπως βλέπετε, έχουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες, όλους τους τομείς, είτε κατά κύριο λόγο, είτε υποστηρικτικό προς άλλους οργανισμούς. Πάνω από 300 αρχές ε, πολιτικές και στρατιωτικές σήμερα έχουν αρμοδιότητα άμεση ή έμεση εκτοφυλακής. Και εμείς ε, τους δίνουμε την προστιθέμενη αξία που χρειάζονται για να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ευθύνες και δραστηριότητες. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων λοιπόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρότεινε και υποστήριξε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ε, την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή τον Ιανουάριο του 2016. Ε, άρχισε και ολοκληρώθηκε στη Λισαβόνα τον περασμένο Ιούνιο στην ΕΜΣΑ ε, με παρουσία και εκπροσώπηση και το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα έχει ένα set test για τη συνεργασία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα στα πλαίσια των μέτρων για την προστασία των συνόρων. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η εγκάσια ε, ε, διακλαδική σημασία των ε, τριών οργανισμών που ασχολούνται με τη φύλαξη των συνόρων και των θαλασσίων συνόρων, Frontex, EMSA και άλλα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα και λειτουργίες ακτοφυλακή. Οι τρει διευθυντέ τώρα δοχεύουμε στο να σα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα στις τρεις αρμόδιες επιτροπές, ε, Τραν, Μπάτζ και Λίμπε, ε, κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Τον Νοέμβριο λέει το αρχικό σχέδιο. Είχε ένα προπαιδευτικό ρόλο λοιπόν και προπαρασκευαστικό αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Οι τρεις οργανισμοί έχουν ε, δημιουργήσει ένα μηχανισμό συντονισμού έτσι ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα διαρευνώντας τις συνέργειες, για το ε, καλό και προς όφελος εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών που έχουν καθήκοντα ακτοφυλακής. Από το 2018 το πρόγραμμα εργασίας των τριών οργανισμών θα έχει ένα κοινό κείμενο που θα τονίζει τις προτεραιότητες για το εκάστοτε έτος πάντα στα πλαίσια ε, της λειτουργίας ακτοφυλακής. Συγκεκριμένο παράδειγμα συνεργασίας είναι αυτό τον καιρό με ελέγχους αλληλευτικών σκαφών από ένα σκάφος μας στη Μεσόγειο. Πριν από λίγες εβδομάδες άρχισε αυτή η αποστολή από την ΕΦΚΑ. Έχουμε αναπτύξει και νέες υπηρεσίες. Ε, με αεροσκάφη και με μια ευρία γάμα δραστηριοτήτων. Ασφάλεια στην ναυσιπλοεία, έρευνα και διάσωση, ε, προστασία των συνόρων, ε, έλεγχη σε σκάφη, σε αλλιευτικά, ακόμα και επιβολή του νόμου στη θάλασσα. Όλα αυτά είναι καθοδόν, είναι ένα νέο μοντέλο για πολιτικές αρχές των κρατών μελών και άλλους θεσμούς τη στιγμή που το κανονιστικό πλαίσιο ε, θα ε, οριστεί για την χρήση μη επαδρομένων αεροσκαφών, drones. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη της ε, υπηρεσίας drones, ιδιαίτερα γιατί πρέπει να έχουμε πάρα πολλούς αισθητήρε σε ένα σχετικά μικρό αεροσκάφος για να ελέγχουμε και να μετράμε ό,τι χρειάζεται. Πάντως αυτό το καιρό έχουμε αυτή την καινοτόμα υπηρεσία και το περασμένο Μάιο στην Ισπανία έγινε και μια επίδειξη. Έχουμε και ένα μικρό βίντεο για να δείτε τι υπηρεσίες παρέχουν τα drone μας. Κατά Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Project financed by the European Parliament to stimulate the cooperation between three agencies to work better in the field of Coast Guard. This is a new initiative which I think is very important and one of our tasks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 εδώ είναι καταπολέμηση λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Um, Και άλλο παράδειγμα, ε, μεταφόρτωσης από μεγαλύτερο σκάφος σε μικρότερο λαθρέων εμπορευμάτων. Και εδώ είναι η καταπολέμηση πετρελοκυλίδας. Then there is solar issue, safety of life at sea, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Άνθρωπος στη θάλασσα. And then, uh, lastly, uh, fisheries control detection. Και τέλος έλεγχος και παρακολούθηση της αληφτικής δραστηριότητας. Aquí lo que tenemos nosotros que podemos las coordenadas, pero solamente to demonstrate what kind of έτσι για να δείτε ενδεικτικά και μόνο τη ροή πληροφοριών που συλλέγουμε ε, καθημερινά από τα drones, ήδη από σήμερα. Okay, then we can continue Λοιπόν, συνεχίζουμε τις διαφάνειες και προχωρούμε στην επόμενη. Έχουμε το σύστημα θέτης που δίνουμε στις αρμόδιες αρχές τις δυνατότητες και τα εργαλεία για να προχωρούν σε ε, ελέγχους στη θάλασσα από 600 αρχές σε όλα τα κράτη-μέλη έγιναν αυτές οι νέοψίες. Υπάρχει ε, ε, εγωμένη οδηγία για το θείο και για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και αυτό σημαίνει 10.000 επιθεωρήσεις ετησίως. Πριν από πέντε εβδομάδες, στις 7 Αυγούστου, επίσης αναπτύξαμε συστήματα στο πλαίσιο θέτης κατόπιν αιτήματο της Γενικής διεύθυνση Κλίμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα θα επιτρέψει στις αρμόδιε εταιρείε. που ε, των σκαφών που καταπλέουν ε, σε ευρωπαϊκούς λιμένες να ε, δηλώνουν τις εκπομπές ρήπων και να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και επαληθεύσεις από τον Ιανουάριο του 2018 έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων των θερμοκηπίου ε, στην αυτιλία γιατί όλα αυτά τα στοιχεία θα δημοσιεύονται και θα ενημερώνονται ετησίως. Αυτό το σύστημα MRV ε, θα επιτρέψει στις εταιρείες να συνεργάζονται με εντεταλμένους επιθεωρητές έτσι ώστε να βελτιώνουν ε, τις επιδόσεις ε, των σκαφών και να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετησίως θα δημοσιεύει συγκεντρωμένα συνολικά στοιχεία ανασκάφους, κατανάλωση καυσίμου, εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και ενεργειακή απόδοση δείκτης κατά μέσο όρο. Μεταξύ άλλων στοιχείων, για πρώτη φορά έχουμε ένα σύστημα που μπορεί ο κλάδος να συλλέγει στοιχεία και να τα ε, διαβιβάζει ε, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε σκάφους. Έρχομαι τώρα στην κρίση του προσφυγικού. Ε, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και μια τρίτη άσκηση ε, στην Νορβηγία ε, για ε, το προσφυγικό. Εδώ συνεργάζονται διάφοροι ενδιαφερόμενοι, ανταλλάσσουν πρακτικές και εμπειρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες ΕΖΕΣ, η βιομηχανία και άλλοι θα κάνουν μια άσκηση προσωμείωσης προσωμείωση ενός ατυχήματος για να δούμε πώς προχωρούν στη διάσωση ε, σε θέματα ασφαλείας και περιβαλλοντικά. Οι επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές εκπονήθηκαν με βάση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα των ε, προηγουμένων δύο ασκήσεων και το έχουμε υποβάλει ως έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτρόπης στο Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Επίσης, προχωρούμε σε ένα ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιας κυκλοφορίας χωρίς σύνορα. Συνεχίζουμε τη διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς υποστηρίζουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα με 8 κράτη-μέλη και τη βιομηχανία, το κλάδο δηλαδή που συμμετέχει, για να ε, δοκιμάσουμε ε, ε, το ηλεκτρονικό μανιφέστο για ένα πρωτότυπο για μια ενιαία θηρίδα έτσι ώστε να έχουμε μια γενική περιφερειακή προσέγγιση όταν πρόκειται για ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τα σκάφη. Αυτή είναι μια διαδικασία δυστυχώ χρονοβόρα, βήμα-βήμα ε, προχωράει. Ακόμα και σήμερα η ναυτιλία έχει τεράστιο γραφειοκρατικό άχθο. Χρειάζονται πολλές φορές διπλές αναφορές, πράγμα που οδηγεί σε καθυστερήσει και χρονοτριβές. Ένα κλάδο που είναι πάρα πολύ διεθνή και εξαρτάται πολύ από τους χρόνους ε, παράδοση. Έχουμε τώρα στην ε, ε, επιχείρηση Κοπέρνικος με δορυφορικές φωτογραφίες ε, που βοηθάει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται δραστηριότητες στη θάλασσα. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά εφαρμογών από εγκεκριμένους χρήστες, θέματα τελωνιακά, επιπολής του νόμου, παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ε, και άλλα. Είναι ε, επιχειρήσεις και υπηρεσίες παρακολούθησης και τηλεπισκόπησης για να κατανοήσουμε καλύτερα το θαλάσσιο το την εικόνα δηλαδή που επικρατεί στη θάλασσα. Μετά το 2020 θα ενταθεί αυτό το πρόγραμμα Κοπέρνικος και θα χαιρόμαστε πολύ να μας υποστηρίξετε για να διατηρηθεί η προσοχή που αφιερώνεται στη θάλασσα. Ο οργανισμός μας εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ε, υποστηρίζοντας ε, τις ε, παραθαλάσσιες χώρες από τη ρήπανση από το πετρέλαιο ή από τα σκάφη. Σε 17 είναι οι κίνδυνοι που έχουμε εντοπίσει ε, και μέσα σε 24 ώρες μπορούμε να βοηθήσουμε με δύο τρόπους, δύο ειδών υπηρεσίες. Ε, στέλνουμε προσωπικό και ε, υλικοτεχνικό εξοπλισμό ε, σε σύγκριση με τον περασμένο Ιανουάριο. Έχουμε αυξήσει το υλικό. Ε, στη Ραβένα σταθμεύουν αυτά στην Αδριατική, στην Ιταλία ε, και ε, έχουμε και δύο σκάφη αντιμετώπισης πετρελοκυλίδων, ένα στη Μάχη και ένα στη Βόρεια Θάλασσα μάλλον και ένα στη Βαλτική. Συγκεντρώνουμε το ενδιαφέρον παγκοσμίω. Η εντολή μα ήδη καλύπτει την υποστήριξη τεχνική βοήθεια στι χώρε τη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ε, έτσι ώστε να αυξηθεί ασφάλεια, ενεργειακή, η παθητική και η προστασία του περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τακτικά και αποστολές από τρίτες χώρες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την μοναδική και συνεργατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων ιδιαίτερα στο περιβάλλον, πράγμα το οποίο αναγνωρίζει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τελευταία της γνωμοδότηση για το ενιαίο προγραμματικό έγγραφο της ΕΜΖΑ, όπου καταγράφει ρητά είναι ελκυστικέ ε, στι χώρε όλου του κόσμου οι δραστηριότητε ε, τη ΕΜΖΑ και προσελκύουν το ενδιαφέρον σε διάφορου πρακτικού και θεωρητικού τομεί. Και εν τέλει θα ήθελα να υπογραμμίσω την αξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση της υπηρεσίας με ολίγα λόγια για την αξιολόγηση αυτή του 2016-2017, μια συνολική αξιολόγηση πολύ θετική, καθώς αναγνωρίζει ότι η ΕΜΣΑ συμβάλλει σε ασφαλέστερο και πιο καλής ποιότητας θαλάσσιο περιβάλλον, με μεγαλύτερη δυνατότητα προλήψης από πλευράς των κρατών μελών και ανταπόκριση σε σημαντικά προβλήματα και κυρίως σε σχέση με την ρήπανση του περιβάλλοντος. Έχουμε μια έκθεση λοιπόν, την έκθεση αυτή αξιολόγησης, την οποία διαθέτουμε και στον ιστότοπό μας και αντίστοιχα θα ε, υιοθετηθεί από το Διοικητικό μας Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017 το σύνολο των συστάσεων που την ακολουθούν. Τώρα περνούμε στην πρακτική εφαρμογή κατόπιν αυτή τη αξιολόγηση και σα ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σα, κυρίες και κύριοι. Είμαι στη θέση σα για οποιαδήποτε ερώτηση. Σα σας ευχαριστώ κύριε Μιλή για την ε, τοποθέτηση, για την παρουσίαση. Πολλά τα θέματα, είτε περιβάλλον, είτε τεχνικά, είτε και διεθνείς πτυχές που μας εκθέσατε. Και πριν δώσω το λόγο στο συντονιστή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κύριο Βίμ Καμπ, θα ήθελα να καλωσορίσω την ομάδα επισκεπτών που έχει προσκαλέσει ο κύριος Φανενκάμπ. Καλώς ήρθατε, είστε εργαζόμενοι στον τομέα των σιδηροδρομικών, ε, στελέχη ε, και λοιπά λοιπές υπηρεσίες των σιδηροδρόμων. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή των Μεταφορών εκ μέρους της ίδιας της Προέδρου της Επιτροπής. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. με σοβαρά θέματα. Παρουσιάζεται μεγάλη κινητικότητα στον χώρο των θαλασσίων μεταφορών. Έχουμε σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έω και 80% των, των ε, εμπορευματικών μεταφορών μέσα τη θάλασσα, Όλο και περισσότερες και οι γεωπολιτικέ, γεωστρατηγικές ε, συνέπειες, ο αντίκτυπος και βεβαίω πρέπει να δούμε το δικό μα μερίδιο, το ευρωπαϊκό μερίδιο, πώ μπορεί να ενισχυθεί. Είδαμε τα μη επανδρομένα αεροπλάνα, τα οποία κάποια στιγμή θα ανήκουν στο παρελθόν και θα πρέπει, μια και ταχύτατα αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι τεχνολογικέ δυνατότητε να προσαρμοζόμαστε διαρκώ. Ο κύριος Φαντανκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τη ομάδα μου θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μιλή για ε, τον επαναδιορισμό του και καλή επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικός ο οργανισμός σας, θαυμαστός. Όπως βλέπετε εγώ είμαι μόνος μου εδώ, οι ε, συνάδελφοι από Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα επιστρέφουν στα σπίτια τους για να δουν πώς λειτουργεί η έμσα στην πράξη στις χώρες τους Εγώ ε, μπορεί να μιλάω εδώ, εκείνοι έχουν εκδηλώσει τις χώρες τους αύριο βέβαια και εγώ προφανώς έχω, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, θέλω να μάθω κάτι για το τι γίνεται στην πράξη ε, με την ε, διάσωση ετούντων άσυλο. Εσείς τους βγάζετε από τα πλοία, τους διασώζετε. Η Frontex το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει, κάποια άλλη υπηρεσία τα σκάφη σας ενέχονται σε αυτή την υπόθεση. Γιατί στα χαρτιά είναι όλα πολύ ωραία και καλά, αλλά ο κόσμος υποφέρει. Και τι κάνει η ΕΜΣΑ, ουσιαστικά τι πάνε από το δικό του χέρι του οργανισμού σας. Να δούμε λίγο και τη συνεργασία επίσης θα ήθελα με τις υπηρεσίες της Βόρειας Αφρικής. Ε, συνεργάζεται με το λιμενικό ε, του Μαρόκου, την ακτοφυλακή, το πολεμικό ναυτικό. Με τη Λιβύη μαθαίνουμε ότι στηρίζουμε την ακτοφυλακή και η Ιταλία τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κατάσταση αυτή. Και τώρα τι βλέπουμε τελευταία, να συγκρούονται ε, δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού ή το, της ακτοφυλακής με μήκυο τύπου γιατροί χωρίς σύνορα στη θάλασσα για τη διάσωση. Τι γίνεται τώρα με αυτό. Θα αφήνουμε τον κόσμο να πνίγεται. Από την άλλη δεν θέλουμε να τους δώσουμε και ένα εισιτήριο για άμεση και απευθείας υποδοχή στην Ευρώπη. Αυτά για το άσυλο. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα, το περιβάλλον. Τα είπατε κι εσείς ότι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και την παγκόσμια διαχείριση διακυβέρνηση των ωκεανών. Σας ρωτώ, στη Μεσόγειο έχουμε αυτή τη σούπα με τις πλαστικές σακούλες, γιατί στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό έχουμε ένα χυλό από πλαστικές σακούλες που επιπλέει τι ε, πρόβλημα έχουμε στη Βαλτική, ε, στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Θάλασσα και ποιος είναι ο μεγαλύτερος ρηπαίνων. Είναι τα σκάφη ή πηγαίνουν εκεί οι κατάλοιπα από απόβλητα από τη στεριά και καταλήγουν στους ωκεανούς. Ο κύριος Μιλή είναι και διπλωμάτης βέβαια άνθρωπος και μίλησε για την ενιαία θηρίδα ε, για τη θάλασσα και εκφραστήκατε με πολύ διπλωματική γλώσσα ε, ότι γνωρίζει μεγάλη προσοχή και ελπίζω να προχωρήσει. Καμία σχέση. Είμαστε σε πολύ κακιά ε, μοίρα και κατάσταση. Πολλέ χώρες και δικιά μου, οι κάτω χώρες, δείχνουν ε, εγωισμούς εθνικούς. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι πιστικό αυτό το προϊόν, αυτή η θηρίδα. Υπάρχουν εθνικές αρμοδιότητες που μπαίνουν εκεί, ξέρω εγώ, αστυνομία, τελωνία, όπου τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ διστακτικά για να μην πω εθνικιστικά και εγωιστικά. Αλλά η ευρωπαϊκή ενιαία ναυτιλιακή θαλάσσια ε, θηρίδα είναι σημαντικό. Σήμερα το πρωί συζητούσαμε για το CITS ε, που δεν καταφέρει να απογειωθεί αυτό το πρόγραμμα. Έρχομαι τώρα στον Κοπέρνικο, αν κατάλαβα καλά. Ε, το είπατε κι εσείς, καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημοφιλής περισσότερο εκτός των τυχών παρά εντός των τυχών. Κοιτάξτε τις σχέσεις σας και τις επαφές με τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες εκτός της Ενώσεως. Είναι λίγο απογοητευτικό να διαπιστώνουμε τι συμβαίνει εντός. Αλλά ας το προχωρήσουμε όμως γιατί είναι και ένα εξογωγικό προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αυτά τα ολίγα και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαντενικάμπε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μάισνερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ εκ μέρου των φιλελευθέρων να σα ευχαριστήσω για την παρουσίασή σα, Είναι λυπηρό το ότι είμαστε τόσο λίγοι εδώ, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μα είπατε. Συναρπαστικά. Έχω και εγώ μια-δυο ερωτήσει. Θα προσπαθήσω να μην διατυπώσω τι ίδιε με τον Βιμ Φανενκάμπ. Κάμπ. Φαντάζομαι βέβαια ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε αντίστοιχε ιδέε στα διάφορα θέματα. Για την ακτοφυλακή και του πρόσφυγε, δεν θα κάνω την ερώτησή μου, μια και έχει διατυπώσει αρκετέ ήδη Βήμα. Για τα μη επανδρομένα όμω αεροσκάφη, τα οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν χρησιμοποιούνται εδώ και, ε, παρά μόνο εδώ και λίγο χρόνο. Ε, πώς ελήφθη αυτή η απόφαση και έχουν ε, αναλάβει έχει ξεκινήσει δραστηριότητα αυτή των μη επαδρομένων αεροπλάνων κατόπιν εντολής ε, των κρατών μελών ε, και βέβαια ποιος πληρώνει το κόστος της χρήσης τους. Για την ε, υποστήριξη των ιοψιών. Από τον Άρθρο του 2017 είπατε μόνο ότι έχει ξεκινήσει ή υπάρχει πιο πολύ καιρό. Ανεξάρτητος όμως του πότε ξεκίνησε, είπετε ότι υπάρχει οδηγία για τις ε, εγκαταστάσεις ε, υποδοχής, τους λιμένες. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί και από την ε, Γερμανία ξέρουμε ότι έχουμε στη Βαλτική σε ένα βαθμό πολλά ζητήματα σχετικά με την εξκαφή των ε, βυθών στους ε, λιμένες με αποδέσμευση σημαντικών ποσοτήτων θείου και αυτό μπορεί να οδηγήσει βέβαια σε, σοβαρές, ε, σε σοβαρή ρήπανση. Μπορεί να το δει αυτό από ψηλά από τον ουρανό με τα συστήματά της η ΕΜΖΑ ή γίνεται κάποιος άλλος, με κάποιον άλλο τρόπο ο έλεγχος των συνεπειών της βυθοκόρησης. Και επίσης, μιλάτε για μια διαδικασία μικρών βημάτων, όντως. Ωστόσο, όταν μιλάτε για double reporting, για διπλή αναφορά, για διπλές καταγραφές, ε, οι επικαλύψεις προκαλούνται από τις ε, ε, διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κάποιο άλλο πλέγμα αυτές οι διπλές, οι επικαλύψεις αναφορών. Είναι το single, το single bundling θα έπρεπε να απλωστεύει τα πράγματα και όχι να τα καθιστά πιο περίπλοκα. Για δε τον Κοπέρνικο που επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, άλλωστε μας παρουσιάσατε και στην ε, παρουσίασή σας έναν κατάλογο προϊόντων. Τι είδου προϊόντα μπορεί να έχει το Κοπέρνικο ε, και τι είναι αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ κυρία Κίλλονεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Γενικό Διευθυντή για την παρουσίασή του και βεβαίως να τον συγχαρώ και εγώ από τη δική μου πλευρά και από την φιλανδική αντιπροσωπεία για την εκλογή του. Σας ευχόμαστε ε, καλή επιτυχία στην, στο δύσκολο έργο σας. Ε, ένα ερώτημα το οποίο συχνά ε, τριβελίζει το μικρό μου κεφάλι όταν συναντάω και συναδέλφους από άλλες χώρες μέλη και όταν ε, γίνεται λόγος για, για τις δραστηριότητες της ΕΦΣΑ, της ΕΜΣΑ, συγγνώμη, αναρωτιόμαστε πόσες επικαλύψεις υπάρχουν στις δραστηριότητες της ΕΜΣΑ σε σχέση με τα όσα γίνονται από τις χώρες μέλη, ε, τα ε, χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καν οι χώρες μέλη πριν προχωρήσουν σε αυτές τις δραστηριότητες να έρθουν σε επαφή με εσά. Και αυτή είναι επικάλυψη. Σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε με σωστό και ευφύ τρόπο τα, τα, τους πόρους μας. Ο κύριος Keith Taylor, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ορισμένες ερωτήσεις να σας κάνω. Πρώτον, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Αυτό δεν ήταν η ερώτηση όμως. Τώρα θα έρθει η πρώτη μου ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας. Πρόλαβα και το ρώτησα εγώ στην κυρία Μέσνερ. Δεύτερον, δεν ξέρω εάν γνωρίζετε, λίγες ε, Κυριακές πριν ε, υπήρξε ένα τοξικό νέφος το οποίο προέρχεται από τη θάλασσα ε, νότιες ακτές της Αγγλίας 150 από τους ε, πολίτες ε, της ε, περιφέρειάς μου πήγαν σε μια όμορφη μέρα και πήγαν στη θάλασσα και έξω γενικά να περπατήσουν αλλά εμφανίστηκε αυτό το τοξικό νέφος και τελικά κατέληξε η ωραία βόλτα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, με μετούς και ζαλάδες. Σας ρωτώ λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε έτσι ώστε να μάθουμε ε, τι προκάλεσε και τι είδους ε, ήταν αυτό το νέφος και εν πάση περιπτώσει ποιος είναι υπεύθυνο για αυτή την έκκληση του νέφους, του τοξικού. Τρίτον, ίσως εκτός θέματος. Αλλά φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποφασίσει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς έχετε προβλέψει κάτι για την περίπτωση που και τη στιγμή που θα συμβεί αυτό το Brexit. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιθ Τέιλορ, λέει η Πρόεδρος. Είναι ένα ζήτημα αυτό ε, το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την την, ε, ε, ε, την Επιτροπή μας η ασφάλεια των θαλασσών και το Brexit είναι δύο θέματα που μας απασχολούν πολύ. Η Αγγλία είναι, Μεγάλη Βρετανία είναι μέλος της υπηρεσίας ΕΜΣΑ. Επομένως η αποχώρησή της θα έχει και δημοσιονομική επίπτωση ε, και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί για τα επόμενα χρόνια. Ερώτηση λοιπόν, έχετε ήδη προβλέψει κάτι έχετε προβλέψει κάτι για να αντισταθμίσετε τις ε, επιπτώσεις, τις δημοσιονομικές ε, του Brexit στην υπηρεσία σας. Όσον αφορά επίσης ε, και τα ε, θαλάσσια ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν αυτά καθεαυτά τη θάλασσα, δεν ε, αναφερθήκατε τι θα γίνει με τα πορθμία, με τα φέρις, τα οποία ε, λειτουργούν σε ενωσιακές περιοχές. τρίτων και εξίσου σημαντικό, ο θαλάσσιος τομέας, ο ναυτικός τομέας ε, έχει μέλλον και θα είναι επίκεντρο προσοχής για τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα 20 χρόνια, ας πούμε, έχετε κάνει κάποια πρόβλεψη πώς θα λειτουργήσουν οι θάλασσες, πώς θα ε, λειτουργεί η οικονομία της θάλασσας, ε, πώς θα λειτουργούν οι ναυτικές και θαλάσσιες αρχές. Έχετε έτσι κάποια πρόβλεψη για ή ένα προσχέδιο απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Thank um, Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι όλες οι ερωτήσεις πολύ ενδιαφέρουσες και καλές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω επάξια. Με τον κύριο Φάντεν Κάμπ ξεκινώ για τους ετούντες άσυλο και πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική που περνούν την Μεσόγειο. Κατά κύριο λόγο. Η δική μας εμπλοκή ε, συνίσταται στο να προσφέρουμε στην ε, Frontex πληροφορίες για ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα. Δηλαδή προσπαθούμε να ε, δούμε μικρά σκάφη που βρίσκονται στη θάλασσα και να διαθέσουμε, να αποστείλουμε στη Frontex τα στοιχεία. Και από εκεί και πέρα ε, έχουν την ευθύνη τα κράτη Frontex να αντιδράσουν στις ε, καταστάσεις αυτές. Δεν είναι δική μας δουλειά, δηλαδή η ΕΜΣΑ δεν παρεμβαίνει, μόνο διοχετεύει τις πληροφορίες. Τις οποίες λέγει με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία που δεν διαθέτουν πάντοτε οι Frontex, οι εθνικές αρχές. Δηλαδή, ο εξοπλισμό υψηλή τεχνολογία δεν είναι πάντα διαθέσιμος. Και αρκετέ ήταν οι περιπτώσεις όπου τα εργαλεία ε, παρατήρησης της ΕΜΖΑ απεδείχθησαν πολύ χρήσιμα για τις αρχές και βοήθησαν να σωθούν πολλές ζωές. Όχι πάντα βεβαίως, γιατί είχαμε και πνιγμούς. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε με τον εξοπλισμό που έχουμε στη θέση μας. Και αντίστοιχα αναπτύσσουμε και την υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε ε, μέσω των μη επανδρομένων αεροσκαφών, μεγάλων επανδρομένων αεροσκαφών που όμως αυτή τη στιγμή παράγονται μόνο για ε, στρατιωτικές χρήσεις με πολύ ψηλό κόστος. Δεν είμαστε σε θέση ακόμη να αγοράσουμε ένα τέτοιο ε, σκάφος, αεροσκάφος, μη επανδρομένο το οποίο θα μπορούσε να διανύσει πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ε, αλλά συνομιλούμε με τους παρέχοντες στη σχετική υπηρεσία και διερευνούμε την κατάσταση. Έχουμε λοιπόν και με τις άλλες υπηρεσίες συνεργασία, ε, όπως και με τις εθνικές αρχές, τις ιταλικές, τις ελληνικές, τις ισπανικές, τις γαλλικές, που έχουν στη συνέχεια και την ευθύνη να ε, αναλάβουν δράση στα διάφορα περιστατικά που τους ε, γνωστοποιούμε. Στη Μεσόγειο έχει αρμοδιότητες ε, σε ορισμένα σημεία το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό, οπότε τους προσφέρουμε τις σχετικές πληροφορίες, όπως άλλωστε και η αποστολή Αταλάντη για, την, ε, για το κέρας της Αφρικής λαμβάνει εκεί την υποστήριξή μας. Και επίσης συνεργαζόμαστε με χώρες της Βόρειας Αφρικής. Εδώ και χρόνια με το SafeMed 3 που έχει ολοκληρωθεί ως πρόγραμμα και τώρα προχωράμε στο SafeMed 4. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας άλλη μια τετραετία με 4 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή μας για την ενίσχυση του δυναμικού των εθνικών αρχών των αφρικανικών κρατών προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια, την, ε, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ε, την εποπτεία των θαλασσών και πάντοτε είμαι στη θέσή τους για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα και σε επίπεδο ισοδυνάμω με αυτό προσφέρεται στις χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Αγωθής της Μεσογείου. Η Γενική Διευθυνσία είναι αυτή η οποία έχει χορηγήσει την παράταση αυτών των εργασιών και τη σχετική επέκταση της χρηματοδότησης. Βεβαίως χώρες όπως από το Μαρόκο μέχρι και την Ιορδανία, από την νότια πλευρά οχθή της Μεσογείου, επίσης με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό συμμετέχουν στο πρόγραμμα γιατί βλέπουν ότι έχουν σαφές όφελος. Και βέβαια έχουμε και πολύ συγκεκριμένε επιχειρησιακές δραστηριότητες ε, με προσφορά από πλευράς μας προς την Τινησία επί παραδείγματι εξοπλισμού που για μας ήταν σχετικά πεπαλαιωμένος, ωστόσο μετά, την, ε, μετά τον εξυγχρονισμό του, τους τον δωρήσαμε και τον εγκατέστησαν στα ε, σκάφη τους προκειμένου να αναπτύσσουν μόνοι τους δραστηριότητες παρακολούθησης της θαλάσσιας ρήπανσης. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα με τα οποία, στα οποία αναπτύσσουμε δραστηριότητες με τις χώρες της νότιας οχθής της Μεσογείου. Ένα θέμα που βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό των πλαστικών ρήπων ε, και γενικά των ρήπων που μας απασχολεί όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και σε όλα στις θάλασσες ε, λόγω των ε, ερμάτων που ανοίγουν τα πλοία και μπορεί να μολύνουν έτσι τις θάλασσες. Η ΕΜΣ αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα όμως. Μπορεί αργότερα να αναπτυχθεί ένα τομέα αρμοδιότητας που σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα μας επιτρέπει να ε, αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο της ρήπανσης από πλαστικά υλικά ε, στις θάλασσες αλλά βέβαια και στις παράκτιες ε, περιοχές η οδηγία για τι εγκαταστάσει υποδοχής πλοίων στους λιμένες ε, είναι μια οδηγία στην οποία συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ένα σύστημα να αναπτύξουμε με το ΦΕΤΙΣ EU, e ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την ε, καταγραφή των ε, δραστηριοτήτων κάθε κάθε σκάφους και πάνω απ' όλα τι είδους υλικό έχει φορτωμένο, τι είδους ε, απόβλητα εγκαταλείπει στον ε, λιμένο. Όπως είπατε όμως τα απόβλητα είναι υπαρκτά ήδη και δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι την ανάπτυξη του προγράμματος θέτης για να τα ε, αντιμετωπίσουμε. Ήδη λοιπόν έχουμε ξεκινήσει να τα αντιμετωπίσουμε, έχουν γίνει κάποιες πρώτες δοκιμές. Ε, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά, αυτό τον εξοπλισμό που λέγεται πλαστικοφάγος, που εγκαθίσταται δηλαδή σε ορισμένα σημεία της θάλασσας και μπορεί να ρουφήξει το πλαστικό υλικό και να το εξαφανίσει. Ε, πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως έχει το σύστημα που μειώνει το διοικητικό φόρτο με την καταγραφή ε, και τις δηλώσεις έπρεπε να είναι λειτουργικό ήδη. Πάμε μέχρι την υλοποίηση των προδιαγραφών των, της οδηγίας από τα κράτη-μέλη που πρέπει να έχει γίνει από το 2015 ήδη. Ωστόσο, ε, η μονοθυριδική προσέγγιση που απαιτείται ε, δεν επιτρέπει επικοινωνία με άλλες αντίστοιχες θηρίδες στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και έτσι δεν έχει ε, φέρει καλά αποτελέσματα αυτό το σύστημα και γι' αυτό ζητούμε αυτή το μονοθυριδικό σύστημα να αναπτυχθεί με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επικληρωθεί μόνο σε 7 ή 8 κράτη-μέλη και περιμένουμε μια πρώτη αξιολόγηση που θα οδηγήσει σε εκτίμηση των ε, αναγκών για αναθεώρηση στην οδηγία, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μονοθυριδικό σύστημα. Αυτό βέβαια σημαίνει συνεργασία και με τα τελωνία και με, τον, ε, με τη βιομηχανία με όλο τον τομέα των θελάσσιων μεταφορών καλύτερα, ε, προκειμένου να δούμε πώς μπορεί το, ε, η φορτωτική του πλοίου να εντάσσεται με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία μέσα σε ένα σύστημα μία και μόνο φορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σύστημα που ξεκινάει το 2016 και έχει περίοδο προσαρμογής έως το 2020. Ξέρετε ότι μπορεί κάποια κράτη να μην έχουν προχωρήσει αρκετά γρήγορα στην ενσωμάτωση των εθνικών του συστημάτων, δεδομένου δε ότι και εμείς δεν έχουμε τρόπο να τα πιέσουμε ή να τα πείσουμε να το πράξουν. Κύριε Μπορώ να κάνω μια μικρή συμπληρωματική ερώτηση. Έχουμε και την αξιολόγηση της οδηγίας 2000 10, ε, 65. Τι διαβάσαμε. Αλλά έχουμε τα πληρώματα τους πλοιάρχους και τις πλειοκτήτριες εταιρείε που διαμαρτύρονται για όλο αυτό το γραφειοκρατικό βάρος που ε, ε, επήλθε χωρίς βελτίωση. Εμείς πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό. Γιατί μπορεί ο καθένας να έχει το σύστημά του, αλλά αν δεν συνεργάζονται κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Exactly, that is Μα ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι. Πρέπει να δούμε πώς δουλεύουν τα συστήματα, πώς ε, συναντιούνται, πώς επικοινωνούν τα συστήματα. Και βέβαια το πλήρωμα που είναι πάνω στο σκάφος ε, πρέπει να τροφοδοτεί μέσα σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ε, στοιχεία τα οποία έχει επί χάρτου. Αυτή είναι η περιπλοκή. Και είπαμε ότι είχαν ε, βεβαίως πληρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη οι προϋποθέσεις της οδηγίας με το μονοθυριδικό σύστημα, αλλά με διαφορετικά συστήματα το κάθε κράτος και άρα το κάθε κράτος μπορούσε να έχει για τους, ε, ειδικά σε αυτά τα κράτη που είχαν μεγάλα ε, λιμάνια, ε, σπουδαία λιμάνια, ε, είχαν δικό του σύστημα και έτσι δεν θέλανε να ενταχθούν σε ένα διαφορετικό. Μία επανδρομένα αεροσκάφη για την κυρία Μάισνερ. Ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα των drones. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια ευρεία παλέτα υπηρεσιών. Μέχρι το 2020 έχουμε δεσμεύσει 67 εκατομμύρια ευρώ για τη δουλειά αυτή. Προχωρούμε σε διάφορους διαγωνισμούς για παρόχους υπηρεσιών και για ταυτοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που χρειαζόμαστε για να ε, εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μας. Ε, ωστόσο, όπως είπα, τα μη επανδρομένα αεροσκάφια που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ σχετικά μικρά. Προσπαθούμε με διαφορετικού τύπου δέκτες να βελτιώσουμε την δυνατότητα ε, συλλογής πληροφοριών και παρατήρησης αυτών των αεροσκαφών είναι μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά πάντως προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σε υπερχόμενες υπηρεσίες. Έχουμε 15 κράτη-μέλη ήδη στο Συμβούλιο μας που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, δηλαδή την κάλυψη των υφισταμένων ε, και των παρεχομένων από την έμψη υπηρεσιών και τη συμπλήρωσή του με, Το θέμα που μας απασχολεί ωστόσο είναι ότι η άδεια πτήσεω πρέπει να προέρχεται από τις εθνικές υπηρεσίες. Ε, δεν μπορεί να χορηγήσει άδεια πτήσεω η ίδια η ΕΜΣΑ, άρα σε κάθε εθνικό ενέριο χώρο πρέπει κάθε κράτο να χορηγήσει τις, ε, τις σχετικές άδειες ε, πτήσεις. Πρώτη μας ε, παρέσχε τη σχετική άδεια πτήσεις η Κροατία και είναι και η πρώτη η οποία υποφελείται από αυτές τις υπηρεσίες για τις οποίες δεν χρειάζεται να πληρώνουν τα κράτη αυτή τη στιγμή που είναι δοκιμαστικό το σύστημα. Είναι δωρεάν όπως και να έχει παροχή αυτών των υπηρεσιών και εν ευθέτω χρόνο θα έχουμε ενδεχομένω και άλλους ε, ενδιαφερομένους ε, υπηρεσίες αεροπορίας που θα χορηγήσουν άδειες πτήσεις σε άλλους εθνικούς ενέργειους χώρους και έτσι θα ενισχυθεί το σύστημα και θα εμπλουτιστεί. Το θείο. Το θείο και, στις, και στους θαλάσσιους όγκους αλλά και στην ατμόσφαιρα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θείο, επί παραδείγματι, στην ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να το μυρίσει το ε, μη επανδρομένο αεροσκάφος. Όταν ε, πετάει πίσω από ένα άλλο σκάφος μπορεί να μυρίσει το καύσιμο που καταναλώνει το αεροσκάφος αυτό και να καταγράψει αν υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. Βέβαια στις θάλασσες είναι πολύ πιο περίπλοκη αυτή η ανείχνευση. Δεν έχουμε δηλαδή εργαλεία για παρακολούθηση διαφόρων τύπων ε, ρήπανσης στις θάλασσες τέτοιου, τέτοιου χαρακτήρα και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμεθα και από τις εθνικές αρχές που θα αποστείλουν ε, σκάφη για να πάρουν δείγμα από μια συγκεκριμένη περιοχή. Δορυφορική όμω δυνατότητα παρακολούθησης της παρου... η ανείχνευση παρουσία θείου στο... στα θαλάσσια ύδατα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνουμε. Ε, μονοθυριδική προσέγγιση και οι διπλές ε, εκθέσεις. Το είπαμε αυτό, ότι είναι ένα πρόβλημα λόγω απουσίας της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών. Πρέπει να τους ασκηθεί πίεση έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα μια στενότερη συνεργασίας και μεταξύ τους. Ε, Κοπέρνικος και οι υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα. Έχουμε προχωρήσει σε ε, συνεργασία με την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση για τον Κοπέρνικο με 40 εκατομμύρια στο 2020 αρχική συμφωνία, χρήματα με τα οποία μπορούμε να ε, συμπληρώσουμε το υφιστάμενο δυναμικό μας σε η απεικόνηση με τη δορυφορική απεικόνηση του Κοπέρνικου. Και έχουμε μέχρι τώρα μία μορφή εικόνας δορυφορικής που όμως δεν είναι ε, άμεση εικόνα, είναι αντικατοπτρισμός. Τώρα όμως μπορούμε σιγά σιγά να... η αντανάκλαση. Τώρα μπορούμε όμως σιγά σιγά να προχωρήσουμε σε ε, άμεση οπτική απεικόνηση. Επίσης συνεργαζόμαστε με ανώτερες σχολές των κρατών. Ενημερώνουμε για τις πρωτοβουλίες μας. Ενημερώνουμε ότι όλα τα ερευνητικά, ε, όλο το ερευνητικό μας προϊόν ε, με το που επαληθεύεται, επικυρώνεται, είναι διαθέσιμο στον ιστότυπό μας. Ο κύριος Τέιλορ μας ε, ρώτησε για ενημέρωση και πληροφορίες, είναι στη διάθεση σας βεβαίως και η παρουσίασή μας. Μία περίπτωση ρήπανσης που αναφέρθηκε για τις... Ε, για ε, το, τοξική ομίχλη, τοξική αχλή, ε, όπως σας είπα μόνο σε σχέση με το θείο μπορεί να ανοιχνευθεί η ρήπανση στον ατμοσφαιρικό αέρα χάρη στους, ε, στα μία παδρομένα αεροσκάφη ε, που μπορούν να μυρίσουν το θείο. Για άλλα όμως ε, τοξικά δεν έχουμε δυνατότητες. Υπάρχουν περιορισμοί ούτως ή άλλως τεχνικού χαρακτήρα σε, αυτούς τους, σε αυτά τα drones, στα μία παδρομένα αεροσκάφη, ίσως μπορέσουμε να τα ενισχύσουμε και ταυτόχρονα όταν θα έχουμε εξασφαλίσει την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθήκων ε, και μέσω δορυφόρου μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτό το επίπεδο. Και το Brexit. Παρακολουθούμε τις συστήσεις των Βρεξελών. Δεν συμμετέχουμε στις συνομιλίες για το Brexit, δεν είναι ρόλος μας αυτός. Βεβαίως και ανησυχούν πολύ, γιατί έχουμε 16 Βρετανούς στην υπηρεσία μας που δεν ξέρουν τι τους επιφυλάσσει στο μέλλον. Ε, ανεπίσημα έχουμε συνομιλήσει με τις Βρετανικές Αρχές βεβαίως και τον αντίστοιχο θαλάσσιο ε, κλάδο, τον κλάδο των θαλασσών μεταφορών της Βρετανίας. Βεβαίως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από την η προοπτική αυτή, γιατί λαμβάνουν πολλές πληροφορίες από εμά χρήσιμες και για τους θαλάσσιους πόρους και ταυτόχρονα ε, και εμείς θα έχουμε πρόβλημα, γιατί και το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει, ή σφέρει στα δικά μας συστήματα πληροφοριών ε, το υλικό του. Άρα ασφαλώς θα έχουμε δυσμενείς συνέπειες από το Brexit στην ασφάλεια την περιβαλλοντική και λοιπή στις θάλασσές μας. Επί Έχουμε στο Αμπερδίν ένα σχετικό αποθηκευτικό χώρο που μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ε, ναυτικών ατυχημάτων ε, και που με τον Brexit θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να μετατοπιστεί ή αν θα χρειαστεί να βρεθεί μια ειδική συμφωνία. Όπως είπα, δεν συμμετέχουμε συζήτηση για τον Brexit, αλλά μπορεί να αλλάξουν αρκετά πράγματα με τον Brexit. Ε, σε σχέση με τα δικά μας θέματα πάντως ε, για τους Βρετανούς, το Brexit θα φέρει την υποχρέωση να αλλάξουν ολόκληρο το σύστημα και το πλέγμα το ρομποθετικό για τη, για τη θάλασσα, για την ε, ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών και την, την, παρακολούθηση της θαλάσσης ρήπανσης και αυτό θα σημάνει τεράστιο όγκο εργασιών και για αυτούς. Αλλά όλα αυτά, όπως είπα, είναι θέματα τα οποία θα κρυθούν στη συνέχεια με τη μορφή που θα πάρει η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να δούμε τι θα γίνει μετά από μια εικοσαετία. Οι θαλάσσιες λεωφόροι λεγόμενες ε, και η ανάπτυξη. Φυσικά θα παραμείνει η ναυτιλία και θα αυξηθεί και υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που θα βρουν νέες λύσεις όμως με ταχύτερους ή βραδύτερους ρυθμούς προχωρούμε. Επίσης ζητούμε όλο και περισσότερο για ε, παρακολούθηση της ναυτιλίας και έλεγχο εξ αποστάσεως, ιδιαίτερα μακρισμένες ε, αποστάσεις. Όλα αυτά ε, είναι θέμα διεθνούς ανάπτυξης. Ε, στα χωρικά ύδατα. Τώρα στην Νορβηγία γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά οι εθνικές αρχές είναι αυτές που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση. των πλήρωμάτων για ε, έλεγχο της ναυσιπλοείας εξ αποστάσεως. Δεν ξέρω, θα χρειαστούν τώρα 20 χρόνια, 25, αλλά προς τα εκεί εδεύουμε έτσι έχει η κατάσταση. Η κυρία Μάισνερ, μια μικρή τελευταία ερώτηση, μάλιστα. Να τα πω γλυκά για να τα καταλάβετε απευθείας. Κάτι που δεν απαντήθηκε ως ερώτημα. Σας ρώτησα τι γίνεται με αυτό τον κατάλογο προϊόντων του Κοπέρνικου. Τι πουλάει ο Κοπέρνικος θα ε, συμπεριλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα που έχετε συλλέξει και μια ερώτηση καινούρια. Γιατί ρώτησε ο Keith Taylor για το Brexit και με την Νορβηγία τι γίνεται. Βλέπουμε τι συμβαίνει στις νορβηγικές ακτές. Ε, εσείς λοιπόν που τα παρακολουθείτε αυτά και έχετε τα στοιχεία, τα διαβιβάζετε στους Νορβηγούς, ακόμα και αν είναι κρατος μέλος. Ε, Μάλιστα, ευχαριστώ για αυτή τη συμπληρωματική ερώτηση. Ο κατάλογος του Κοπέρνικου συμπεριλαμβάνει όλες τις ε, υπηρεσίες που παρέχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εμπεριστατωμένη εξήγηση και συνολική των δυνατοτήτων και των ε, καθηκόντων μας. Θα ακολουθήσει και νέος. Δεν θέλω τώρα να σας ε, προεξοφλήσω το καινούριο κατάλογο θα έχετε πρόσβαση και ήδη για το σημερινό έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας να δείτε ποιες είναι οι υπηρεσίες. Η Νορβηγία είναι χώρα ΕΟΧ. ΕΖΕΣ μάλλον. Έχουν τις ίδιες ε, δυνατότητες, ελέγχουμε την ακτογραμμή τους, ε, συνεργαζόμαστε. Για μας είναι σαν ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Είπα, voilà. Να λοιπόν ε, τελείωσε εδώ το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά που μας ε, απαντήσατε, που μας παρουσιάσετε τις προκλήσεις ε, του Οργανισμού Ασφάλειας στη Θάλασσα. Στην αρχή και μόνο βρισκόμαστε, στις ψηφιοποίησεις των νέων εξελίξεων. Σήμερα το πρωί μιλούσαμε για αυτοκίνητα με αυτόνομη οδήγηση. υπάρχουν ε, και τα πλοία χωρίς ε, ε, πλήρωμα. Επίσης υπάρχει μετανάστευση, μετακινήσεις πληθυσμών, θα δούμε και νέους πρόσφυγες να φτάνουν στις ακτές μας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, και είναι πάρα πολύ πολύτιμος ο ρόλος σας. Αλλά φυσικά το πιο σημαντικό είναι η οικονομική υποστήριξη. Είπατε ότι το προσωπικό σας ανησυχεί η Βρετανοί, αλλά έχουμε ευρωπαϊκές αποστολές ε, πέρα από τους Βρετανούς. Ε, θα πρέπει όλες οι χώρες να υποστηρίζουν, να βοηθούν τον οργανισμό σας, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στο πλευρό μας και πάντα μπορούμε να υπολογίζουμε στη βοήθειά σας για να προχωρούμε από κοινού. Δεν το βάζουμε κάτω. Είναι μεγάλα τα προβλήματα. Το πρωί ζήτησαμε τη διακυβέρνηση των ωκεανών και εκεί μεγάλες προκλήσεις για ένα καλύτερο πλανήτη, αλλά και ε, για να υπάρχουν οι θάλασσες μας και αύριο. Αυτά. Λήξη συνεδρίασης. Θυμίζω, συνάδελφοι, ότι θα τα ξαναπούμε στις 25 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Το σημειώσατε όλοι, 20 27 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα και αν δεν έχετε άλλη αντίρρηση, κυρίως το πέρα συνεδρίες και